Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε για να προχωρήσουμε με την συνεδρίασή μας. Το τελευταίο σημείο που έχουμε στη σημερινή ημερήσια διάταξη έχει να κάνει με τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Καταρχάς θα ακούσουμε μία παρουσίαση για τις ε, δραστηριότητες και για το ιστορικό του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας και μετά στα μέλη της Επιτροπής θα δοθεί ευκαιρία να επισκεφθούν το, τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας και βεβαίως θα δείτε και ένα βιντεάκι σχετικά. Τον Μάιο του 2017 ε, έγιναν ε, τα εγγένεια της, ε, του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και βεβαίως η Επιτροπή παρακολουθεί από την αρχή αυτή την δραστηριότητα. Έχουν γίνει πολλές επισκέψεις στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας από μέλη της Επιτροπής μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω την κυρία Ιτσελ και τον κύριο Ντουκ που είναι εκπρόσωποι του οίκου και ήρθαν σήμερα εδώ να μας παρουσιάσουν κάποια στοιχεία. Θα σας δώσω τώρα το λόγο. Θα σας δώσω 15 λεπτά και στους δύο. Οπότε, όποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτος μπορεί να το πράξει. Σας ακούμε. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής σας. Είναι βεβαίως ε, μεγάλη τιμή για εμένα ως ε, Γενικού Διευθυντή ε, για, για την επικοινωνία να είμαι προσκεκλημένο σήμερα εδώ. Ξέρω ότι είσαστε ιδιαίτερα απασχολημένοι. Είναι οι πρώτε εβδομάδε άλλωστε τη καινούργια μάλλον θητεία του Κοινοβουλίου και γι' αυτό πραγματικά είναι μεγάλη χαρά και τιμή και για μένα και για την ομάδα μου να είμαι εδώ σήμερα για να σα παρουσιάσω τον οίκο τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Μα με συνοδεύει ο διευθυντή Σίριλ Στόκελη και όπω είπατε και εσεί, η Διευθύντρια του οίκου Ευρωπαϊκή ιστορία, η Κωνστάνσε Ιτσελ. Και βεβαίω ε, είναι κάποια μέλη και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου εδώ μαζί μα. Η δουλειά σα ε, ε, στην Επιτροπή σα συνδυάζεται με, τα όσα με τα όσα κάνει η δική μας Γενική Διεύθυνση. Ε, πραγματικά νομίζω ότι όλοι είμαστε παθιασμένοι με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, όχι αφηρημένα, αλλά σε πολύ συγκεκριμένε δραστηριότητες της ε, κοινωνία μας μέσω πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να μπορέσουμε να ε, προωθήσουμε τα προγράμματα Εράσμους αλλά και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού έτους ε, κληρονομιά, όσο πιο πολύ προς τους πολίτες μας. Ξέρετε ότι κάτω από την ε, Γενική Διεύθυνση της, ε, για τις Επικοινωνιών έχουμε ξεκινήσει διάφορε δραστηριότητε και έχουμε πολλέ εγκαταστάσει εδώ για του επισκέπτε, εδώ στι Βρυξέλλες και βεβαίω κάποιε και σε κράτη-μέλη. Αυτέ οι εγκαταστάσεις έχουν στόχο να υπογραμμίσουν τη δουλειά που γίνεται και στι χώρε σα και στι εκλογικέ σα περιφέρειες, δίνοντα χώρου όπου οι πολίτε μπορούν να έρθουν και να μάθουν για την Ευρώπη και μπορούν βεβαίως να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο που παίζει η Ευρώπη στη ζωή μας. Ο οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι η τελευταία άφηξη. Είναι ας πούμε ο νέος μαθητής στην τάξη στις εγκαταστάσεις που έχουμε εδώ για τους επισκέπτες της Βρυξέλλες από την ε, μέρα που άνοιξε για το κοινό το 2017 το μουσείο αυτό έχει εδραιώσει τη θέση του και ως κομμάτι των εγκαταστάσεων για τους επισκέπτες του Κοινοβουλίου. Ε, αποκινούμε το ημικύκλιο και το Παρλαμεντάριο που είναι το κέντρο των επισκεπτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ως ένα σημείο που πρέπει κανείς να δει ε, ως τουρίστας στο Βέλγιο, και μάλιστα τώρα είναι, ε, βρίσκεται στη δέκατη θέση ε, όσων ε, αξιοθέατων πρέπει να επισκεφθεί κάποιο όταν έρχεται στι Βρυξέλλε, το TripAdvisor. Ο λόγο πίσω από την επιτυχία του νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα μουσείο το οποίο δεν το έφτιαξαν οι διοικητικοί υπάλληλοι, δεν το έφτιαξαν οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου, το έφτιαξαν άνθρωποι που ε, ασχολούνται με, την, ε, με τα μουσεία και ιστορικοί. Ε, δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να έχουν πολύ υψηλή ποιότητα επισκέψεις. Η επίσκεψη μπορεί να γίνει και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι μπορούν οι επισκέπτες να παρακολουθούν τις εκθέσεις στη δική τους μητρική γλώσσα και με την ταχύτητα που τους διευκολύνει και επίση οι επισκέπτες ε, νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας ε, μπορούν να ε, σκεφτούν με έναν τρόπο κριτικό και ει βάθος για την ιστορία της Υπήρου μα και για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τους ε, προπάτορες μέχρι το Brexit, από το ε, παρελθόν ε, μέχρι τις σημερινές διαδηλώσεις. Έχουμε μάλιστα και μια, ένα κομμάτι αφιερωμένο στο μουσείο για τις διαδηλώσεις που γίνονται για την αλλαγή του κλίματος. Ε, θα καταλάβετε λοιπόν ότι το μουσείο αυτό είναι ένα μέρος που εξελίσσεται. Είναι μια δουλειά που α, εναλλάσσεται συνεχώς. Όπως βεβαίως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. το μουσείο αυτό ε, προσπαθεί να έχει πολλές δραστηριότητε ε, και να αποτελεί ένα μέρος ανταλλαγή απόψεων, συζήτησης και εδώ στις Βρυξέλλες επιτόπου αλλά και στο διαδίκτυο. Και μάλιστα έχει δημιουργήσει και ένα ε, εκτεταμένο πρόγραμμα εκμάθησης για επισκέψεις ε, από σχολεία. Όταν θέσαμε αυτούς τους ε, ε, φιλόδοξους στόχους, ε, ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας, αλλά βεβαίως και η δική μου Γενική Διεύθυνση, θέλουμε να υποστηρίξουμε και τη δική σας την δουλειά ως εκλεγμένων προσώπων του, των Ευρωπαίων πολιτών και θέλουμε βεβαίως να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τι πολιτιστικέ και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Κωνσταντσε Ίτσελ, που είναι η επικεφαλή, η διευθύντρια του Οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας, αλλά πριν από αυτό νομίζω ότι υπάρχει και ένα πολύ σύντομο βιντεάκι, το οποίο θα δούμε, θα σα παρουσιάσει τον Οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία, το μουσείο μα, και βεβαίω θα σα εξοικειώσει και εσά με το τι κάνουμε και τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Και στο τέλος αυτής της παρουσίασης και τη δική μου και τη Κωνσταντσε, Ευχαριστώ να σα απαντήσουμε και σε ερωτήσει, αν έχετε. Σα ευχαριστώ.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 shaped by traditions, sustained by people. Here is our story. Yes, uh, dear members of the uh, Committee on Culture and Education. Αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή Πολιτισμού, θέλουμε να σα δείξουμε αυτό το σύντομο φιλμάκι για όσου δεν μπορέσουν να προβούν στην επισκέψη σήμερα. Να σε ευχαριστήσω στο όνομα όλη τη ομάδα μου για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω αυτό το μουσείο. Από τότε που αρχίσαμε να εργαζόμαστε γύρω στο Νίκο, η Ευρωπαϊκή Ιστορία στο 2008, έχουμε έρθει τουλάχιστον μια φορά του χρόνου στην Επιτροπή, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις ό,τι αφορά το μουσείο αυτό. Το οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία είναι το πρώτο μουσείο που δείχνει την ιστορία από μια προοπτική ευρωπαϊκή, διεθνική και βεβαίω συνδυάζει στοιχεία από τοπικά, περιφερειακά και εθνικά μουσεία. Έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και έχουμε φτάσει στι 300.000 επισκέψει πριν από μερικέ μέρε. Έχει μεγάλη, μεγάλη επιτυχία το μουσείο. Έχουν, αυξάνονται οι επισκέπτε, είναι πολύ καλέ οι κριτικέ και είναι πολύ υψηλό το ποσοστό ικανοποίηση. Φέτο λάβαμε ε, μία, ένα βραβείο από το Ευρωπαϊκό Μουσείο, για το Ευρωπαϊκό Μουσείο του Χρόνου που αναγνωρίζει ότι το, η ο οίκο Ευρωπαϊκή ιστορίας ε, δημιουργεί ευαισθητοποίηση για την σημασία των ευρωδημοκρατικών αξιών, τα ανθρώπινων δικαιώματα και την ποικιλομορφία. Είναι ένα νέο κέντρο για την κριτική ανάλυση ευρωπαϊκή ιστορία και ένα φόρουμ για την αναζήτηση και την ε, εξερεύνηση των παρόντων πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων. Το μουσείο έχει γίνει ένα σοβαρό εταίρο για καθηγητέ ιστορία, ε, μουσεία, λόγω της ακαδημαϊκής του ανεξαρτησία και, τη, και της επαγγελματικότητας σε, σε μουσιολογικό επίπεδο. Υπάρχει μια ακαδημαϊκή επιτροπή και ένα ε, διοικητικό συμβούλιο τον οποίο ε, ο πρόεδρός σας και άλλο ένα μέλος είναι μέλη de facto. Θα ήθελα να αναφερθώ σε στοιχεία που δεν θα δείτε στη σημερινή έκθεση. Θα επικεντρωθώ λοιπόν μόνο στις δραστηριότητε μας ό,τι αφορά τις συλλογές τις εκδηλώσεις και τις ε, δραστηριότητες επικοινωνίας και εκμάθησης. Σε ό,τι αφορά τις συλλογές τώρα, όπως είδατε στην ταινία, οι εκθέσεις βασίζονται κυρίως σε δάνεια, αλλά η αποστολή είναι να συλλέξουμε και στοιχεία και έγγραφα, ντοκουμέντα, τα οποία δεν έχουν συλλέξει εθνικά και περιφερειακά μουσεία. Αυτά συνδέονται με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προκατόχων της. Κανένα άλλο μουσείο στην Ευρώπη για την ώρα δεν επικεντρώνεται σε αυτή την ιστορία. Ο οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία λοιπόν θεωρεί ότι είναι δική του αποστολή να προστατεύσει αυτή τη κληρονομιά. Τώρα το πρόγραμμα εκδηλώσεων. Πέρα από τις προσωρινές και μόνιμες ε, εκθέσεις, ε, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε σε μεγάλες εκδηλώσεις όπως το, ε, τη Μέρα Κληρονομιάς, οι νυχτερινές επισκέψεις σε μουσείο, και συζητούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις για μια σειρά αποζητήματα. Φέτος, παραδείγματο χάρη, μιλήσαμε το 1989. Αυτό ήταν το θέμα προς συζήτηση. Συχνά ε, συνδέονται αυτέ οι εκδηλώσεις με τις προσωρινέ εκθέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, πολύ σημαντικέ προβολές που έχουν να κάνουν με την προσωρινή έκθεση Restless Youth και στι νυχτερινές μας ε, παρουσιάζουμε και έργα νέων σχεδιαστών μόδας και αυτό αποτελεί, συνδέεται και με την έκθεση. Τώρα τα προγράμματα εκμάθησης, αυτά έχουν να κάνουν διάφορες, ε, έχουν διάφορες ομάδες στόχους, ε, ηλικιωμένους, οικογένειες, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ε, ο στόχος είναι ε, να οργανώσουμε ε, tour με οδηγούς, ε, ημέρες για την οικογένεια, άλλες δραστηριότητε και βεβαίως τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε 24 γλώσσες Εσεί είστε υπεύθυνοι για τα ζητήματα εκπαίδευση σε αυτήν την επιτροπή. Καλό είναι να γνωρίζετε λοιπόν ότι κάνουμε και κατάρτιση καθηγητών για το περιεχόμενο ε, των εκθέσεών μα. Έχουμε πάνω από 100 ε, πόρου online, τα, οι οποίε είναι δωρεάν προς, ε, ε, για να τα κατεβάσουν, εν περιπτώσει, στο διαδίκτυο. Θέλουμε να συνεισφέρουμε για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της ιστορίας. Τέλος, έχουμε κάποιες δραστηριότητε επικοινωνίας. Είναι το μόνο στον κόσμο που έχει μια ιστοσελίδα σε 24 γλώσσες στο μουσείο μας. Έχουμε και διάβλους με τα κοινωνικά, κοινωνικούς, κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Όπως συμβαίνει με τα μουσεία, ε, δημοσιεύουμε ε, βιβλία για την ιστορία, καταλόγους των εκθέσεων. Έχουμε γράψει και ένα βιβλίο για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το ειδικό μουσείο ε, μπορούμε να στο, στο στείλουμε αυτό, διότι είναι αρκετά έτσι ογκώδες, μια διεθνής ομάδα ιστορικών σε 24 γλώσσες, σε ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, προτίμας αυτό το μουσείο, είναι κάτι το μοναδικό. Καλό είναι να γνωρίζετε ε, ότι έχουμε δημιουργήσει και μια υπηρεσία VIP που είναι στη διάθεσή σας για τις ομάδες ψηλού επίπεδου. Θέλουμε επίσης να σας καλέσουμε επισήμω να, να στέλνετε τι ομάδε επισκεπτών σα στο, στον οίκο μα, διότι αυτό το μουσείο είναι το μόνο μουσείο ιστορίας όπου μπορεί κανεί να μάθει από τι εμπειρίε από την Ανατολή, τον Νότο, το Βορρά, την Δύση τη Ευρώπη ε, Μπορούμε πολλά να μάθουμε δηλαδή από τις εμπειρίε άλλων. Κλείνοντας, κάποια σχόλια για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δύο χρόνια μετά τα εγγένεια, το μουσείο έχει αναπτύξει μια σειρά από πολιτικές για να αναπτύξει περαιτέρω μια σειρά από δραστηριότητε. Έχουμε καθορίσει ένα πρόγραμμα προσωρινών εκθέσεων για τα επόμενα τρία χρόνια και βεβαίω αναπτύσσουμε συνεχώ και δοκιμάζουμε και αξιολογούμε τα προγράμματα κατάρτιση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε όλο και πιο ευρείε ομάδε στόχου. Εξετάζουμε ποιοι έρχονται στο μουσείο, ποιοι δεν έρχονται, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την προσφορά μα έτσι ώστε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερου ανθρώπου. Όπω δείχνουν οι μελέτε των επισκεπτών μα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ε, επισκεπτών από την Δυτική και Νότια Ευρώπη. Θέλουμε να βρούμε τρόπο να βγούμε από τους τοίχου του μουσείου. Έχουμε ψηφιακά project όπω ε, ένα, εικονικό, ε, ένα εικονικό tour του μουσείου. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τι λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί για να βελτιώσουμε την προσφορά μα προ του επισκέπτε. Ελπίζω να βρείτε τον το χρόνο να μα επισκεφτείτε τη σήμερα το απόγευμα ή κάποια άλλη στιγμή και βεβαίω είμαι στη διάθεσή για να απαντήσω στα ερωτήματά σα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ιτσέλ. Ευχαριστούμε κύριε Ντούκ για την ε, παρουσίασή σας. Καταρχάς να ρωτήσω αν θέλουν οι συντονιστές το λόγο. Αν θέλετε, ευχαρίστως να σας ακούσουμε. Η κυρία Κάμεραβερτ, Πέτρα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχάς, ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και που μας καλέσατε να επισκεφθούμε το μουσείο. Θέλω να είμαι σύντομη για να δώσω το λόγο στους, να δώσω τη δυνατότητα στους νέους συναδέλφους να θέσουν ερωτήματα. Εγώ απλώς θέλω να πω ευχαριστώ, γιατί εν τω μεταξύ έχω στείλει πολλές ομάδες και έχω προσκαλέσει πολλές ομάδες επισκεπτών να πάνε στο μουσείο και νομίζω ότι όλοι όσοι πήγανε κάθε φορά ενθουσιάζονταν από την αρχή δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχε πάει τόσο καλά αυτό το project, ότι η ευρωπαϊκή ιστορία δηλαδή θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα τόσο μικρό χώρο, γιατί το μουσείο δεν είναι τεράστιο, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά ως προς αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει πολλά, έχει εξελιχθεί πολύ το μουσείο και πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ και από εδώ και μπρος επίσης καλή επιτυχία. Εγώ σίγουρα θα συνεχίσω να στέλνω τους επισκέπτες μου στο Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε και εσείς Τη δραστηριότητα σα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζωηντόβα. Ε, Ευχαριστώ πολύ και την Διευθύντρια και τον ε, Διευθυντή. Έχω έρθει πολλές φορές ε, στο μουσείο και πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερο την εργασία σας. Στην αρχή της προηγούμενης χρονιάς οργανώσαμε ε, ε, παρουσίαση ενός ε, ντοκιμαντέρ, ενός φιλμ για τον Κάλλας, γιατί είχε, ήταν η, η επέτειος της... Αυτοκτονίας του. Και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ερώτηση. Υπάρχουν στατιστικές για τους ε, φοιτητές ε, ή τέλος πάντων για τις ομάδες ε, των, τις κατηγορίες των επισκεπτών. Θα με ενδιέφερε να καταλάβω πώς είναι οι επισκέπτες και σε ανακατηγορία πώς είναι. Δεύτερη ερώτηση. Κάποια χρόνια πριν ε, υπήρχαν κάποιοι προβληματισμοί ή φόβοι ότι ίσως δεν θα ήταν πολύ καλή η ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του μουσείου και των ε, εκθέσεων ή ο τρόπος με τον οποίο ε, θα παρουσιαζόταν κάποια πρόσωπα σε αυτήν την στην αφήγηση της ιστορίας. Συμφωνώ ότι το μουσείο είναι ζωντανό και ενεξελίξει διαρκώς ποιες ήταν οι αλλαγές που κάνατε ή ποιες αλλαγές προετοιμάζετε έτσι ώστε να υπάρχει απαραίτητη ισορροπία. Πάντως, να σας πω ότι αξιολογώ πολύ θετικά και εκτιμώ την εργασία σας και ελπίζω ότι και οι καινούργιοι βουλευτές θα, θα επισκεφτούν ε, τον οίκο ε, και θα αποκτήσουν ίδια γνώμη. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ για την εργασία που κάνετε. Βεβαίως έχω επισκεφθεί ήδη το μουσείο, τον Νίκο, αυτό τον Νίκο ε, της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Άλλωστε είμαι ιστορικός, τουλάχιστον αυτό ήταν το πρώτο μου πτυχίο. The history, uh, some months after... Uh, ε, πραγματικά θα ήθελα να ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που αναφέρονται εκεί και να σας πω ότι και στη χώρα μου ε, υπάρχει ομάδα ιστορικών που ε, ήθελε να έχει πρόσβαση ε, στα ιστορικά στοιχεία και πρέπει να πω ότι η ευρωπαϊκή ιστορία ακόμα είναι γραμμένη από την οπτική γωνία της Δυτικής Ευρώπης και αυτό εξηγείται από την ιστορία μας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε ισορροπία, μια δηλαδή γεωπολιτική εξισορρόπηση. Προσπαθείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Έχετε επίσης ε, και ε, πρόθεση από ερευνητική πλευρά. έχετε κάποια στρατηγική ερευνητική έτσι ώστε να επανέλθει αυτή η ισορροπία ε, και να παρουσιάζουμε την ιστορία χωρίς ιδεολογική τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαρό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και τον ε, κύριο Διευθυντή και την Διευθύντρια. Ευχαριστούμε πολύ ε, και για την επίσκεψη που θα μας κάνετε. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά την εκπαίδευση στην ιστορία, γιατί νομίζω ότι αυτά που θα δούμε και η ποιότητα της, της ιστορικής έρευνας είναι πραγματικά δεδομένα. Αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν για το μέλλον. Δηλαδή, ε, κατάλαβα ότι έχετε ε, ήδη επιγραμμικά ε, παιδαγωγικό υλικό. Τα έχετε προωθήσει τα υλικά αυτά στις διάφορες χώρες μέλη γνωρίζουν οι διδάσκοντες ας πούμε ότι υπάρχει το υλικό αυτό δουλεύετε, ας πούμε, συνεργάζεστε με τα Υπουργεία ε, Παιδείας ε, όσον αφορά αυτό το επιγραμμικό υλικό. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ ένα, μια μικρή παύση για να ακούσουμε τις πρώτες απαντήσεις. Oui, euh, Dank, Frau Ευχαριστώ την κυρία Κάμερα για τα πολύ καλά σας λόγια. Να απαντήσω πρώτα στην κυρία Έχουμε στατιστικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά το συσχετισμό μεταξύ ομάδων και ατομικών επισκεπτών. Έχουμε διαπιστώσει με μεγάλη έκπληξη ότι για το έτος 2018, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 50% επισκεπτών κάτω των 30 ετών. Έχουμε δηλαδή πολλούς νέους. Τώρα που θα αναπτύξουμε και μια πολιτική για να απευθυνθούμε σε νέο κοινό θα μελετήσουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό για να καλύψουμε και πιο ε, μεγάλες ηλικιακές ομάδες. Ε, μπορούμε να στείλουμε εξαιρετικά στοιχεία αν σας ενδιαφέρουν για την κατανομή αναχώρα, για το ποιες γλώσσες επιλέγουν πάνω στο τάμπλετ οι επισκέπτες, ε, αλλά δεν θέλω τώρα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή τα αξιολογούμε όλα αυτά το ζήτημα της ισορροπίας. Ε, νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ε, ε εκπόνηση της μόνιμης έκθεσης με όλους τους ε, ενδιαφερόμενους. Βρήκαμε μια συμβαστική λύση, θεωρούμε έτσι βιώσιμη, με βάση την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Τα σχόλια συχνά είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος που σύμφωνα με τους επισκέπτες ή ε, τους ιστορικούς ή τους ε, δημοσιογράφους λείπουν είναι ένας ατελείωτος κατάλογος θα χρειαζόμασταν δεκαπλάσιο χώρο και πάλι δεν θα μας έφτανε πάντως εξετάζουμε ιδιαίτερα το θέμα της ισορροπίας μεταξύ, βορά, μεταξύ Ανατολής και Δύσης ε, και Βορρά και Νότου είμαστε σε μια φάση αξιολόγησης έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές όπου θεωρούσαμε ότι είχε γίνει κάποιο λάθος κάποια λάθος, καθασμένη κρίση εκ μέρους μας αλλά θα κάνουμε και μια αξιολόγηση λίγο πιο σε βάθος μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας, διότι συχνά τα σχολεία είναι τόσο αντιφατικά μεταξύ τους, που είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε τη μία κατεύθυνση σε βάρος της άλλης. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση αξιολόγησης. Νομίζω ότι απάντησα ε, στο ερώτημα της ισορροπίας. Τώρα, θέσατε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για, για μας, γιατί βαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην ιστοριογραφική έρευνα. Βεβαίω από τότε που το 2008 ενέκρινε το, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ε, ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη οδηγία, ε, επειδή έχουμε πολύ συγκεκριμένου πόρου, δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί ίδιοι την έρευνα. Μπορούμε να, τα, να ενθαρρύνουμε ε, ανταλλαγέ μεταξύ ερευνητών από διάφορα μέρη τη Ευρώπη. Το κάνουμε αυτό, παραδείγματο χάρη με αυτήν την σειρά ε, Debating Histories. Ε, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και πόρους ε, που είναι καινούργοι ε, και που έχουμε στη διάθεσή μας μετά την πτώση του τείχους αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι αυτή την έρευνα διότι η δική μας ομάδα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της έκθεσής μας. Είναι πάντως ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μας. Εάν υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο έρευνας ή κενά, αυτό μπορούμε να το καλύψουμε με τις συζητήσεις μεταξύ ιστορικών έτσι ώστε αυτό το πρόβλημα να αναδειχθεί. Τώρα, η εκπαίδευση και η ιστορία. Πολύ σημαντικό το θέμα για, ε, για μας. Αυτό που θα θέλαμε είναι τα μαθήματα ιστορίας να γίνουν λίγο πιο ευρωπαϊκά, λίγο πιο διεθνικά, υπερεθνικά, να, να προσθεθούν στην εθνική ιστορία, διότι διαπιστώσαμε ε, από τους επισκέπτες μας αλλά και από την ομάδα μας ότι η εκπαίδευση συνήθως είναι εθνική, είναι της εθνικής ιστορίας ή και περιφερειακή σε κάποιες χώρες και χρειάζεται να γίνει μια μεγάλη δουλειά για να καταλάβει κανείς την προοπτική του άλλου. Εμείς έχουμε αναπτύξει αυτούς τους πόρους ε, επιγραμμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, σε μια τάξη ας πούμε και όχι μόνο στο μουσείο, αλλά πρέπει να γίνει μεγαλύτερη δουλειά διάδοση αυτών των, των στοιχείων. Συνεργαζόμαστε με το δίκτυο των καθηγητών ιστορίας, ε, Ευρω... Ευρωπαίων καθηγητών ιστορίας, ε, προσπαθούμε ε, να αυξήσουμε τη διάδοση αυτή, έχουμε και τα σχολεία πρέσβης, εάν υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες όπως παραδείγματο χάρη ενημέρωση μέσω των Υπουργείων Παιδεία. Αυτό θα ήταν κάτι που θα μα ενδιαφέρει. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σα. Euh, Ίσως θα μπορούσα να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε και η κυρία Ίτσε προηγουμένως. Ε, δηλαδή εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει ε, τις αρμοδιότητες ε, του οίκου. Βεβαίως η ιστορία μας βοηθάει γιατί έχουμε τη δυνατότητα και επιγραμμικά και με άλλο τρόπο να έχουμε εργαλεία εκπαιδευτικά αλλά γιατί και γιατί μας δίνει και την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με διάφορα φόρα στα οποία μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε στο μέλλον, μάλλον πώς θα οργανωθεί στο μέλλον η διδασκαλία της ιστορίας, είτε πρόκειται εθνική ιστορία, είτε ιστορία των εθνών, είτε ιστορία με κεφαλαίο γιώτα. Ε, επίσης υπάρχει και ένα ε, σχέδιο το οποίο ε, δεν σχετίζεται άμεσα με τον οίκο. Υπάρχει πρόγραμμα συνεργασίας με σχολεία και κάθε χρόνο σε αυτό το πρόγραμμα που ονομάζουμε το πρόγραμμα των πρέσβεων προσθέτουμε διαρκώς ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε περισσότερα σχολεία, σε περισσότερα παιδιά, σε περισσότερες οικογένειες. έτσι ώστε να προσθέσουμε και κάτι στο ορολόγιο πρόγραμμα των παιδιών ε, που διδάσκονται ιστορία στην Ευρώπη. Βεβαίως, ε, οι κυβερνήσεις είτε περιφερειακές είτε εθνικές είναι αυτές ε, που καθορίζουν το πρόγραμμα των σχολείων, πόσες ώρες θα διδαχτούν τι και επομένως είναι δικιά τους αρμοδιότητα και επομένως εμείς κάνουμε περισσότερο δουλειά σε πολιτικό επίπεδο και όχι τόσο σε διοικητικό. Επίσης όσον αφορά τις ισορροπίες, πολλές ισορροπίες υπάρχουν στον οίκο γεωγραφικές και σχεδόν και ιδεολογικές θα τολμούσα να πω στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα στοιχεία. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες ε, όσον αφορά τον τρόπο που η Δυτική Ευρώπη κυρίως έβλεπε ε, την ε, ιστορία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν ποτέ δεν μπορεί κανείς να φτάσει στην ομοφωνία, αλλά νομίζω ότι έχουμε πετύχει το, την καλύτερη δυνατή ε, ισορροπία. Ε, έτσι ώστε τα μηνύματα ε, και το υλικό που παρουσιάζεται να είναι ισορροπημένα. Εγώ είμαι Ισπανός. Κάποια στιγμή ε, συνόδευσα ε, και ομάδες βουλευτών από την Ισπανία ή επισκεπτών από την Ισπανία ε, και υπήρχαν ε, κάποιοι που είπαν ότι για την Ισπανία περισσότερα πράγματα περιέχει ο οίκος από το πιο μαύρο παρελθόν ας πούμε του φασισμού και λοιπά της ιστορίας και όχι από το τι συμβαίνει τώρα ε, και υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι έλεγαν ότι θα έπρεπε με καλύτερο τρόπο και πιο αναλυτικά να παρουσιάζονται ε, οι, ε, ο, το, ο τρόπος με τον οποίο υπέφεραν οι άνθρωποι στην Ισπανία στη δικτατορία. Επομένω, ομοφωνία είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει. Προχωρούμε λοιπόν τώρα. Παρακαλώ ένα λεπτό ο καθένας από εδώ την προς. Κυρία Άντερσον έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Δυστυχώς ε, δεν ε, ε, μπορούσαμε να τα πούμε όλα. Είναι πολύ καλό αυτό που είδαμε στο βίντεο. Μας ανοίγει την όρεξη για περισσότερα. Εγώ σίγουρα θα περάσω να το δω το μουσείο. Είναι και έτσι διαδραστική η δραστηριότητα. Θα με ενδιέφερε εμένα να δω πώς το διαχειρίζεστε, γιατί καμιά φορά οι νέοι δύσκολα ενδιαφέρονται για την ιστορία Έχετε κάποια αίσθηση για το πώς μπορείτε να φέρετε πιο κοντά στους νέους στην ιστορία, δηλαδή έστω και έτσι διαδραστικά ενδιαφέρονται περισσότερο για την ιστορία. Als nächstes ist... Επόμενος, η κυρία Μπούντινγκ. Hello, once again, Oleka. Ναι, ε, σας ευχαριστώ και εγώ για τις παρουσιάσεις και βεβαίως ε, ε, προσβλέπω στην, απο, στην απογευματινή μου ε, επίσκεψη. Για μας που είμαστε καινούργοι, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο ποια είναι η συνεργασία με το Παρλαμεντάριο, γιατί εγώ είδα λίγο την ιστοσελίδα του μουσείου όσο μιλούσατε, είδα κάποιες από τις εκθέσεις, ε, κάποια πράγματα που νόμιζα ότι γίνονται στο, παραλμε, στο Παρλαμεντάριο μου δεν γίνονται, ή τέλος πάντων μπορεί να γίνονται, αλλά ίσως γίνονται και παράλληλα στο μουσείο σας. Δεν ξέρω πώς συνδέονται ακριβώς. Και επίση συμφωνώ με αυτό που είπατε για του νέου που είπε η συνάδελφο τώρα γιατί και στο, παραμελτα... στο Παρλαμεντάριο υπάρχει και αυτή η έκθεση, ε, πώς τη λένε, ακόμα και στα αγγλικά τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, ε, για την επανάσταση, διαφόρων ειδών επαναστάσεις. Ε, τι ακριβώς κάνετε, ε, παίρνετε το, τα όσα αφορούν τους νέους στο δικό σας το μουσείο από το Παρλαμεντάριο, πώς ακριβώς το διαχειρίζεστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τεβέσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ίτσε και τον κύριο Ντούκ για την παρουσία τους αλλά και την παρουσίαση που μας έκαναν. Ε, εγώ προσυπογράφω το ε, σχέδιο αυτό, πραγματικά το γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό και θεωρώ ότι είναι μια ψηφίδα πολύ σημαντική ε, στην προσπάθεια οικοδόμησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας αλλά και σημαντική για τους πολίτες της Ευρώπης. Όμως υπάρχει μια απόφαση, δηλαδή να ξεκινήσει η ιστορία από τη Γαλλική Επανάσταση, πολύ ωραία. Θα μπορούσε όμως κανείς ε, να ε, πιστέψει, να, να ακολουθήσει μάλλον ε, το, τους ιστορικούς που λένε ότι ξεκινάει η ευρωπαϊκή ιστορία από το Μεσαίωνα. Μήπως θα μπορούσε να διευρυνθεί λοιπόν η έκθεση. Δεύτερον, Σαφώς πρόκειται για ευρωπαϊκή ιστορία, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε ακριβώς να μεταφέρουμε την ε, εικόνα αυτής της ευρωπαϊκής ιστορίας. Όμως, ταυτόχρονα, ίσως λείπει η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή η ιστορία της ευρωπαϊκής ιδέας, του ευρωπαϊκού ιδεόδους. Ε, γιατί όντως ξεκινάμε ε, εδώ από την ιστορία της Ευρώπης που ξεκινάει μετά από τον πόλεμο όμως ε, υπάρχει και μια προσπάθεια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που έχει ξεκινήσει πολύ πριν με τον Αριστιδη Μπριάν και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να ενταχθεί με κάποιο τρόπο στο πρόγραμμα του μουσείου, του οίκου. Μια σύνοψη λοιπόν και πάλι και σας δίνω και πάλι το λόγο, παρακαλώ αν μπορείτε εντός των χρονικών ορίων. Λοιπόν, για τους νέους ρωτήσατε. Ναι, είναι πολύ, αποτελούν μεγάλο κομμάτι των γενικώ των επισκεπτών μας. Έχουμε κάνει διάφορες έρευνες για τη χρήση του τάμπλετ, γιατί είναι αρκετά περίεργη συσκευή να χρησιμοποιεί κανείς ένα μουσείο αλλά είδαμε ότι δεν εξαρτάται από την ηλικία το πόσο φιλική στο χρήστη είναι η συσκευή αυτή. Εμείς έχουμε κάνει αρκετά μακροσκελείς ερευνές για το αντίκτυπο που έχει το μουσείο, δηλαδή τι παίρνει μαζί του ο νέος. Οπότε θα έχουμε ε, περισσότερα στοιχεία για το πώς το καταλαβαίνουν, πώς, πώς εξοικειώνονται με το μουσείο οι νέοι. Γιατί τα δεδομένα αυτά, βεβαίως θα είναι ανώνυμα φυσικά, αλλά θα μπορούμε και εμείς να αξιολογήσουμε λίγο περισσότερο τον αντίκτυπο του μουσείου στους νέους. Αλλά γενικώ είναι πολύ δημοφιλές στο μουσείο με τους νέους. Ε, για το Παρλαμεντάριουμ τώρα. Είναι μια ε, συμπληρωματική η συνεργασία που έχουμε. Ε, άνοιξε το 2011 το Παρλαμεντάριουμ. Έχει, μια, έχει ένα μικρό ιστορικό τούνελ, αλλά εμείς πάμε πολύ πιο βαθιά στην ιστορία στο μουσείο, γιατί κυρίως το Παρλαμεντάριουμ εξηγούν το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ εμεί είμαστε ιστορικό μουσείο και ασχολούμαστε με όλη την Ήπειρο, όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους, προδρόμους της. Ε, έχουμε ε, αναλύσεις, ιστορικά έγγραφα, ιστορικά αντικείμενα. Οπότε είναι λίγο διαφορετική η δική μας η ε, παρέμβαση. Και βεβαίως, φυσικά έχουμε πάντα στόχο τους νέους. Κάνουμε εργαστήρια, workshops, διαδραστικά, διαδραστικές δραστηριότητες. Προσπαθούμε να έχουμε έτσι μια ανάμεικτη δραστηριότητα για να μπορούμε να δώσουμε κίνητρο σε όλους τους επισκέπτες. Τώρα για την επιλογή της ε, ιστορίας του 19ου και του 20ου αιώνα. Από την αρχή το μουσείο ήταν ε, μουσείο σύγχρονης ιστορίας. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μιλούσε για την ε, ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 20ο αιώνα, το πρώτο μισό του, Ευρωπαϊκού αιώνα, του 20ου αιώνα, αλλά βεβαίως πάμε και πιο πίσω και στον 19ο αιώνα γιατί εκεί ήδη υπάρχουν ε, επαναστάσεις, υπάρχει εθνικισμός, ε, απεικιοκρατία και αυτά είναι νομίζω σημαντικοί ε, όροι που θα πρέπει να εξηγηθούν. Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και πιο πίσω στην ιστορία. Ε, πάντα όλοι οι, ε, υπεύθυνοι των μουσείων ενοχλούνται όταν δεν μπορούμε να δείξουμε πολύ, πολλά στοιχεία της ιστορίας. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το, ό,τι κάναμε για την ιστορία και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα δείτε και το απόγευμα υπάρχει έτσι ένας μπούσουλας μέσα στην έκθεση. Αλλά επειδή είναι και ο χώρος περιορισμένος πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια επιλογή και είναι πολύ εύθραυστη αυτή η ισορροπία για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο, το όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε και από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και κάποιες προσωρινές βεβαίως ε, εκθέσεις, οπότε έτσι μέσω αυτών μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Το ευρωπαϊκό, ε, το ευρωπαϊκό φυσικά υπάρχει, εννοείται, Έχουμε την, ε, το κίνημα Pan Europa που εκπροσωπείται. Μιλούμε για ε, αντιστασιακά κινήματα. Ε, είναι θέματα που επανέρχονται στις, μέσα στις μόνιμες εκθέσεις μας αυτά. Λοιπόν, και τώρα συνεχίζουμε. Ο κύριος Αντέμοφ έχει το λόγο. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας. Είμαι μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα το μουσείο. Θα το κάνω λοιπόν με μεγάλη χαρά σήμερα. Δεν γνωρίζω τις ε, τον τρόπο λειτουργίας του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας, εξού και το ερώτημά μου. Οργανώνεται εκθέσεις ε, προσωρινές ή που επικεντρώνονται σε κάποιες ιστορικές φιγούρες ε, σημαντικές στην ευρωπαϊκή ιστορία ή όταν έχουμε κάποια επέτειο και ε, έτσι, αν γινόταν κάτι τέτοιο, οι επισκέπτες θα είχαν ε, τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα πράγματα για κάτι που συνέβη μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή μια συγκεκριμένη περίοδο ή για μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Ευχαριστώ. Νίκλας. Νίκλας, ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Θέλω να επανέλθω πριν από το μουσείο αυτό. Αρχικά, είχαμε πει, είχε ψηθεί το θέμα του πώς θα ξεκινήσουν αυτές οι εκθέσεις, από, από πού θα ξεκινήσουν μάλλον. Και εγώ συμφωνώ να ξεκινήσουμε από την αρχή, να πάμε όσο γίνεται πιο πίσω δηλαδή. Διότι έτσι νομίζω μπορεί να είμαστε όλοι πιο ικανοποιημένοι. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να, να εξεταστεί και το, και ο Καρλομάγνος, η εποχή του Καρλομάγνου και το βασιλείο του, γιατί είναι σημαντική η χρονική στιγμή ένα ερώτημα. Υπήρχε αυτή η ιδέα να μην έχουμε έναν οίκο στις Βρυξέλλες. Καλό είναι που υπάρχει βέβαια, αλλά τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καλό είναι που έχουμε τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, αλλά όχι γιατί, γιατί μόνο ένα μουσείο, γιατί μόνο στις Βρυξέλλες, όλα είναι στις Βρυξέλλες. Βεβαίω, όταν κάποιο κάνει μια επίσκεψη στι Βρυξέλλε ω φοιτητή, μπορεί να τα επισκεφθεί όλα μαζί αλλά μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες, περισσότερα σπίτια, περισσότερους οίκους ευρωπαϊκής ιστορίας ή να έχουμε μια κινητή έκθεση. Herr Slavakov, Sie haben das Wort. Здравейте на всички уважаеми. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σαμπάκοφ. Δεν θα μιλήσω και ιδιαίτερα πολιτικός ορθά. Τέθηκε ένα ερώτημα. Γιατί δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες χώρες έχουν ε, προσφέρει περισσότερα στην ευρωπαϊκή ιστορία περισσότερα από άλλα, από άλλες χώρες. Όμως η χριστιανική Ευρώπη είδε το φως γύρω στα 800. Λείπουν εδώ γύρω στα χίλια χρόνια. έχουμε κάνει μια προσπάθεια εδώ και χρόνια να ενώσουμε την Ευρώπη εδώ και αιώνες. Η Βουλγαρία υπήρχε ενώ δεν υπήρχε ακόμα το έθνος Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί λοιπόν μικρές χώρες παραμερίζονται. Είμαστε μια ένωση ισότιμων μελών και πρέπει να επανέλθει η ισορροπία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά, αλλά εγώ είμαι μέλος του κόμματος του Brexit και θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ιστορική στιγμή αυτή, έτσι, διότι πραγματικά θεωρώ ότι το να πάρετε την απόφαση να έχετε έναν στόχο να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο που το έχουν φτιάξει οι επαγγελματίες ε, και ιστορικοί είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Εγώ είμαι ε, φαν του μουσείου αυτού. Δεν θα είμαι σήμερα το απόγευμα γιατί το έχω, έχω πάει πολλές φορές. Μου αρέσει πολύ και το τάμπλετ που υπάρχει. Πραγματικά έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ερώτημα μου είναι το εξή όμως. Εγώ θα, σας, ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ ε, ε, εφόσον έχετε κάποιες κόκκινες γραμμές ευρωπαϊκής ένταξης, οι οποίες όμως δεν πρέπει να φτάσουν στο όριο της προπαγάνδας. Θα πρέπει λοιπόν να αντισταθείτε στις σιρήνες που ακούγονται και από εδώ, ότι πρέπει να γίνει ουσιαστικά μια έκκληση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό είναι προπαγάνδα. Δεν είναι μουσείο, ούτε ακαδημαϊκή ιστορία. Γίνεται ε, πολιτικ, ιστορία. Και εσείς δεν το κάνατε αυτό μέχρι τώρα. Και η μεγάλη επιτυχία είναι ότι αυτή η ιστορία, η ιστορία των ευρωπαϊκών ιδεών είναι η ιστορία των ευρωπαϊκών εθνών ε, και ευρωπαϊκέ ιδέε. Δεν είναι το ίδιο με την ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση όμω. Ό,τι και αν πιστεύει κάποιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ω μουσείο σα παρακαλώ πολύ να μην ακολουθήσετε την οδό τη προπαγάνδα, διότι θα είναι καταστροφή για εσά, για την αξιοπιστία σα, ενώ έχετε ένα υπέροχο μουσείο που έχετε φτιάξει. Wir werden jetzt noch äh, äh, einen Redner aufnehmen. Λοιπόν, ακούσουμε άλλον ένα ομιλητή, τον κύριο Ντέα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, να συγχαρώ όλους όσοι οργάνωσαν αυτό το μουσείο. Ε, είναι πολύ σημαντικό να θυμίζουμε τους μεγάλους πολιτισμούς ε, της Ελλάδας, της Μακεδονίας ε, κλπ Νομίζω ότι η Ευρώπη στην ουσία ξεκινάει με τον Καρλομάγνο. Γεννιέται ε, μετά τον ε, ε, Καρλομάγνο. γιατί από εκεί άρχισαν να οργανώνονται και οι πολλές, αυτοί οι διαφορετικοί πολιτισμοί οι οποίοι ήφαναν εν τέλει την Ευρώπη. Πολύ ωραία τα παρουσιάζετε πάντως και σας συγχαίρω. Ich habe auch noch eine Έχω κι εγώ μια παρατήρηση και ένα κοπλιμέντο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το μουσείο. Είναι πολύ σημαντικό και για τις επόμενες γενιές. Αυτό που μου είπαν όμως είναι ότι κάτι λείπει από το μουσείο ή δεν είναι επαρκές. Η ιστορία των μεγάλων μειονοτήτων στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός να ασχοληθείτε και με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θεωρείται ένας οίκος που μπορεί να αναπτυχθεί. Μπορεί ή θα πρέπει να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Οπότε ρωτώ. Επειδή στην Ευρώπη έχουμε μεγάλη αύξηση του ε, ακροδεξιού λαϊκισμού. Θα πρέπει η ε, πολιτισμική παρέμβαση του μουσείου να είναι λίγο πιο ορατή, πιο εμφανής. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, κάποιο σχέδιο προς αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση. So, to start from the top, um... Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οι, οι ε, προσωρινές ε, εκθέσεις. Όπως θα δείτε και το απόγευμα, οι προσωρινές αυτές εκθέσεις έχουν σχεδιαστεί με εταιρείε που ασχολούνται με την παρουσίαση αυτών. Προσπαθούμε να διαλέγουμε πάντα μεγάλα θέματα, γιατί θέλουμε δυόμιση χρόνια για να τις προετοιμάσουμε. Οπότε δεν μπορούμε να τις περιορίσουμε σε ένα ή λίγα αριθμητικά στοιχεία. Οπότε αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε με τις διάφορες εκδηλώσεις μας. Έχουμε ε, ε, σχέδια που ασχολούνται με το 1989. Έχουμε προγράμματα που είναι ε, παρόντα στις, και στις μόνιμες και στις προσωρινές εκθέσεις μας. Σε αυτές τις μεγάλες εκθέσεις θα είναι δύσκολο να επικεντρωθούμε μόνο σε μία προσωπικότητα ιστορική, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλέ. Τώρα για τις προηγούμενες περιόδους, βεβαίως θα Θέλαμε να πάμε και πιο πίσω στην ιστορία, αλλά το θέμα είναι και τι μπορεί να χωνέψει τελικώ ο επισκέπτης. Ε, ο επισκέπτης έχει ένα φάσμα προσοχής 90 λεπτών. Με βάση αυτό προσπαθήσαμε να οργανώσουμε το μουσείο μας. Δηλαδή τι μπορεί να ε, αποκομίσει ένας άνθρωπος σε 90 λεπτά. Θα δείτε ότι και ο χώρο είναι πολύ περιορισμένο. οπότε έτσι έγινε η επιλογή. Αυτό βεβαίω δεν μα αποτρέπει καθόλου να έχουμε προσωρινέ ε, εκθέσει ή να τις ε, τροποποιούμε. Βεβαίως χρειαζόμαστε πάντα καλή προετοιμασία. Δεν νομίζω ότι έχουμε παραμελήσει ή έχουμε ξεχάσει μικρές χώρες. Εγώ δεν το ερμηνεύω έτσι. Αν μπορούμε να δούμε γιατί από την Βουλγαρία. Έχουμε πολλά αντικείμενα από τη Βουλγαρία σε εκθέσεις. Μπορείτε να το δείτε και από τη βάση δεδομένων μας. Και επίσης μπορούμε να παίξουμε λίγο, μπορούμε να αλλάξουμε τα αντικείμενα. Οπότε αν υπάρξει υπερπαρουσίαση μιας χώρας μπορούμε να έχουμε παράδειγμα ας πούμε επαναστάσεων από μια άλλη χώρα. Οπότε αλλάζουν τα ιστορικά κοιμήλια. Προσπαθούμε πάντα να επιτύχουμε μια ισορροπία. Η ακαδημαϊκή ανεξαρτησία τώρα που αναφέρατε είναι κομμάτι ε, της ηθικής ενός ε, μουσείου. Δεν κάνουμε προπαγάνδα. Είναι κομμάτι του δεντολογικού μας κώδικα αυτό. Έχουμε τη μέθοδο εργασία μας. Μας έχει υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς αυτό σε όλη την ε, εκπόνηση του project και βεβαίως από την ε, προηγούμενη ε, θητεία, από τους προηγούμενους πρόεδρους της Επιτροπής εδώ και χαιρόμαστε που μπορούμε να δουλεύουμε με πολύ υψηλά επαγγελματικά πρότυπα. Τώρα, οι μεγάλοι πολιτισμοί. Το ίδιο ερώτημα με αυτό που έχω απαντήσει μερικώς. Αυτό ίσως θα μπορούσε να μπει σε κάποιο άλλο μουσείο, αν υπάρχει τέτοια πολιτική βούληση. Θα θέλαμε όμως όντως να έχουμε εκθέσεις που να μπορούν να ε, περιδιαβαίνουν ουσιαστικά όλη την Ευρώπη. Αλλά βεβαίως αυτό είναι πάντα θέμα πόρων και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ομάδα των υπευθύνων και στις Βρυξέλλες ή γύρω-γύρω στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μετά, για τους ε, Ρωμά, για το ολοκαύτωμα και, τα πεντα... και το μισό εκατομμύριο θυμάτων που αναφέρονται στην έκθεση. Πρόσφατα κάναμε μία εκδήλωση, κάνουμε και εξωτερικές εκδηλώσεις για το Ευρωπαϊκό ε, βραβείο ε, για τα πολιτικά δικαιώματα, για τους Ρωμά. Έχουμε λοιπόν επαφή με την κοινότητα και μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο μπορούν να γίνουν αλλαγέ στην ε, μόνιμη έκθεση και να ενισχύσουμε το χώρο που έχουμε αφιερώσει σε αυτή τη μειονότητα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Αλλιώ, παρακαλώ, υπενθυμίστε το μου. Εκκρεμεί ένα ερώτημα. Η δυνατότητα ο οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία να μην υπάρχει μόνο στι Βρυξέλλες αλλά και σε άλλες χώρες. Ε, ε, αυτό θα ήταν καταπληκτικό να μπορούσαμε να ε, διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε τα μουσεία από πλευρά όμω οργανωτική και δημοσιονομικής κυρίως ε, δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε αυτό το μειονέκτημα, ότι βρίσκεται δηλαδή μόνο στις Βρυξέλλες ε, το μουσείο. Όπως είπε και η Διευθύντρια, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη δυνατότητα της επίσκεψης online, χρησιμοποιώντα δηλαδή ε, τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, έτσι ώστε να έχει κανείς τη δυνατότητα ε, να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε μέρος αυτών που εκτίθενται στο μουσείο και εξετάζουμε και την δυνατότητα να οργανώσουμε εκθέσεις ε, σε διάφορες χώρες με τη σφραγίδα ποιότητας βέβαια της, ε, του οίκου μας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια με τη συνεργασία των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού στα κράτη-μέλη και βεβαίως θα προσπαθήσουμε επίσης, γνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι θέμα του οίκου, είναι μια άλλη πλατφόρμα διαφορετική, Europa Experience. Θα προσθέσουμε λοιπόν να μεταφέρουμε σε μια σειρά από χώρες ε, μικρές ε, ε μινιατούρες, αν θέλετε, ρέπλικες ε, του Παρλαμεντάριου. Θα γίνει αυτό στην, στην, στην, Εσθονία, στην Εσθονία, στο Βερολίνο υπάρχει εδώ και δύο χρόνια, θα το κάνουμε και σε άλλες χώρες, να υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την υποδομή για να ε, συνδεθούμε με κάποια από τα περιεχόμενα του οίκου. Αυτό που θέλουμε επίσης είναι να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ε, δηλαδή σε κάποιες χώρες να μπορέσουν να ξεκινήσουν προ... παρεμφερείς πρωτοβουλίες ή από μουσεία που υπάρχουν ήδη. Ε, έχουμε λοιπόν μια πολιτική επαφών το προσωπικό δηλαδή του οίκου η ιστορική κτλ. Ε, είναι σε επαφή με ιστορικούς άλλων μουσείων ευρωπαϊκών και κάποιοι άλλοι θεσμοί επίση θα μπορούσαν να αντιγράψουν αυτό το μοντέλο. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματο χάρη, συνεργαζόμαστε με το Αυστριακό Κοινοβούλιο που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποια στιγμή αυτό θα μπορούσε να μα επιτρέψει όχι να έχουμε έναν νίκο ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά ε, παρεμφερεί μοντέλα τα οποία αναπτύσσουν ε, άλλοι θεσμοί σε άλλε χώρε. Τελειώνοντα, ε, θέλω να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τα καλά σα λόγια, για το ενδιαφέρον που δείξατε και για τι κριτικέ σα και για, κυρίως για την υποστήριξη. Το πιο βασικό είναι ότι ο οίκος αυτός ε, θα πρέπει να ε, λαμβάνει την πολιτική υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω όλους όσους μπορέσουν να επισκεφθούν το μουσείο σήμερα και για όσους δεν θα μπορέσουν να σας καλέσω να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Ενημερώστε μας, ε, ειδοποιήστε μας ε, για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε και ένα πρόγραμμα ε, για σας ανάλογα και με το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός ε, ανάμεσα στο Παρλαμεντάριο από τη μία και ε, τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας από την άλλη ναι, ε, και υπάρχει και ένα τμήμα της ε, έκθεσης σήμερα και αύριο που θα επισκεφθούμε. Ο κύριος Αδάμov ρώτησε εάν προετοιμάζουμε εκθέσεις και για συγκεκριμένα ειδικά γεγονότα. Ναι, ας πούμε για την 30η επέτειο της πτώσης του ε, τείχους του Βερολίνου. This is one, only one example that we are focusing within parliamentary... Σε συνεργασία με αντίστοιχο Μουσείο του Βερολίνου. Ε, ναι, και επομένως η απάντηση είναι ναι, ότι θα κάνουμε και θα διοργανώνουμε εκθέσεις ε, για συγκεκριμένα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας. Σας ευχαριστώ αξιότιμοι προσυκλημένοι για την παρουσίασή σας και για τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Καταρχάς, λίγο την προσοχή σας τώρα, συνάδελφοι. Όσοι θέλουν να επισκεφθούν τον οίκο της Ευρωπαϊκής Θεωρίας, παρακαλώ να συγκεντρωθείτε έξω από την αίθουσα σε 10 λεπτά και με τη βοήθεια συναδέλφων από την γραμματεία θα πάτε στο Μουσείο της Ευρωπαϊκής Θεωρίας ιστορίας. Η ακρόαση του κυρίου Γκάμπριελ θα γίνει αύριο το απόγευμα και η επόμενη τακτική μας συνεδρίαση θα γίνει την 1η Οκτωβρίου από τις 3 μέχρι τις 30. Ευχαριστώ όλους. Καλό απόγευμα.